είναι και καθήλυνα αρμόδια. Περνάμε τώρα στι ψηφοφορίε. Έκθεση Λούνατσεκ. Συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωσης Κωσοφοπεδίου. Ενιαία ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Διορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο διορισμός ε, θα γίνει ε, στις υποψηφιότητες από την διάσκεψη των Προέδρων. Δεν έχω λάβει τροπολογίες, ούτε τη για από τη διάσκεψη των Προέδρων. Θεωρούνται λοιπόν οι υποψηφιότητες και προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές. Συμφωνίες σύνδεσης σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εδάφη 26. Προφορική τροπολογία Γκάλερ. Σας παρακαλώ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από τη στιγμή που υπάρχει επιτέλους μια νέα κυβέρνηση στη Μολδαβία πρέπει να ενημερώσουμε το κείμενο. Εγώ συμφώνησα με τον κύριο Φλέξταεν από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Αν δείτε τον κατάλογο ψηφοφοριών του βλέπετε το κείμενο λέει χαιρετίζει τη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αδιεξόδου και προσπαθειών που δεν είχαν καρποφόρηση για τη δημιουργία κυβέρνηση και καταλήγει ζητώντα από τα κόμματα τη Μολδαβία να ενισχύσουν την πολιτική σταθερότητα για να μπορεί να υπάρξει μια επιτυχή περάτωση των μεταρρυθμίσεων και ελπίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα μπορέσει να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Αντιρρήσει για αυτή την τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 26 όπως τροποποιήθηκε προφορικός. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, απορρίφθηκε. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος. Έλεγχο, έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας.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 να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα της παραγράφου 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Παρντών. Πέρας. Απορρίπτεται. Εδάφιο 44. Προφορική τροπολογία του κυρίου Φλέκενστάιν. Σας παρακαλώ κύριε Φλέκενστάιν. Κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε <clears throat> την εξή τροπο, τροποποίηση λαμβάνει υπόψη της τις ε, επικείμενες Ολλανδικές κτλ. Και, και όχι εκφράζει τις βαθιές ανησυχίες τους σε σχέση όχι εκφράσει τι ανησυχίε του, αλλά καταγράφει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν. Υπάρχουν αντιρρήσει για αυτήν την τροπολογία. 40. Είναι 40 όσοι έχουν αντιρρήσει. Δεν είναι 40. Οπότε ψηφίζουμε. Παράγραφος 44 όπω τροποποιήθηκε. Προφορικό. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Τροπολογία 1. Σας παρακαλώ. Για διαδικαστικό θέμα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάνω από 40 όσοι σταθήκαμε όρθιοι και δεν μετρήσατε σωστά. Θέλουμε να ελεγχθεί ο αριθμός. Να με συγχωρείτε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν σαφέστατο Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τη ρήτρα αμοιβαία άμυνα βάσει του άρθρου 42 της συνθήκης. Τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία, συγγνώμη. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 18. Υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη Αι. Αρχικό κείμενο. πέρα. Κατά. εκεί εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη των συνόδων του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Τροπολογία 2. Διανάταση χειρό υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφό 29 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Για τη 18. Για την τροπολογία 2. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 307-320. Αν δεν σηκώνετε όλοι τα χέρια από εδώ, είναι αδύνατο να είμαστε και ακριβέστατοι. Παράγραφος 29 σε δύο τμήματα, διανάταση χειρός, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 38. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Με συγχωρείτε. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Παράγραφος 31. 31 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, διανάταση ισχυρό. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Πρώτο τμήμα. Για να χειρός υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 38, παράγραφος 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 45. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Και πάλι η ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 46. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 86 και πάλι διονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 89. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 8-1. Η τροπολογία διανάταση χειρός υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Ε, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Γκέριγκερ. Ντεόντεμπεργκ. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014. Τροπολογία 11. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα δυνατές ισχυρό, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε γιατί δεν σηκώνω όλα τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δυνατές ισχυρό υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. δυνάτα ισχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται. Αλλά σε ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα. Διανάταση ισχυρός. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ναι, αλλά συνάδελφοι, είναι αδύνατο να καταλαβαίνει κανεί ε, δυνατέ ισχυρός αν δεν σηκώνεται όλα τα χέρια. Θα ελέγξουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Διανάταση ισχυρό υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ωραία λοιπόν, α κάνουμε την επαλήθευση, α κάνουμε τον έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Ε, άμα δεν σηκώνετε τα χέρια, πώ να αποφασίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Διανάταση ισχυρό υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Διανάταση ισχυρό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Διανάταση ισχυρό υπέρ. Με συγχωρείτε, παράγραφος 6. Όχι, τροπολογία 6. Διανάτες ισχυρός υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Είμαστε στην παράγραφο 9 σε δύο τμήματα διανάτας ισχυρός πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία παράγραφος 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 21 σε δύο τμήματα. Δυναμαστικής ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δυναμαστικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα δυναμαστικής ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος. Έλεγχο. Θέλετε έλεγχο. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Καλά το είδαμε. Απορρίφθηκε. 34. Πρώτο τμήμα. Διανάταση χειρό υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 35. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 για την αντιλογική σκέψη ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όμως, όμως δεν σηκώσατε τα χέρια σας όλοι. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ετυλογική σκέψη Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχο. Ας κάνουμε έλεγχο για την ετολική σκέψη Q. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. X, Χ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη A, G σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική ψηφοφορία. έρχεται ψηφοφορία. Εγκρίθηκε.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 Προχωρούμε στις επεξηγήσεις ψήφων βάσει της υπηρεσίας διάταξης. Ξεκινούμε με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδίου. Σύσταση της συναδέλφου της κυρίας Λούνατσεκ. Έχουν ζητήσει το λόγο πρώτη η κυρία Μορβάη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι έλλειψη σεβασμού να αρχίσω να μιλάω κάτω από αυτές τις συνθήκες